πράξεις οι οποίες ε, εγκρίθηκαν με την κανονική νομοθετική διαδικασία, οι τίτλοι των οποίων θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στις εργασίες μας. Έχετε ήδη λάβει το σχέδιο ημερήσια διάταξης. Ε, για τη Δευτέρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Για την ε, Τρίτη έχουμε έτοιμα τη ε, κυρίας Λίχτενβέργκερ για άρση ασυλίας της κυρίας Μόρβαϊ, κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί στις ψηφοφορίες Τρίτης. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε η έκθεση Quist Robolt για την κοινή εμπορική πολιτική, οποία προβλέπεται αυτή τη στιγμή να ψηφιστεί την Τρίτη, να συζητηθεί Τρίτη βράδυ. Θέλει κάποιος τον λόγο. Ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για την έκθεση αυτή δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή κάποια συζήτηση. Πρόκειται για τα ζητήματα όμνιμπους της εμπορικής πολιτικής και κατ' ουσίαν πρόκειται για εφαρμογή των νέων νομοθετικών δικαιωμάτων μας στον τομέα αυτών και θεωρώ σωστό να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια και θα ήθελα την στήριξή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κάσπαρη. Θέλει κάποιος να διαφωνήσει με τον κύριο Κάσπαρη. Ή αν κάποιος άλλος θέλει να υποστηρίξει την πρόταση αυτή. Όχι. Κάποιος εναντίον. Όχι. Οπότε παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι όσοι συμφωνείτε με το αίτημα του κυρίου Κάσπαρη. Κατά. Αποχές. Οπότε η συζήτηση της έκθεσης Κουίστρα ε, Ρόβολτ προστίθεται ως τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει την Τετάρτη. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε δήλωση της ε, ΥΠΑ της εκπροσώπου και αντιπροέδρου για την κατάσταση Λευκορωσία την Τετάρτη μετά τη συζήτηση για την κατάσταση στην Ιγυρία. Παρακαλώ, κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο έχει χειροτερεύσει η κατάσταση στη Λευκορωσία, η πολιτική κρατούμενη στη χώρα αυτή και η κρίση η οποία δημιουργήθηκε με τους Ευρωπαίους πρεσβευτές που συζητήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο απαιτεί να γίνει συζήτηση και στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν παρακαλώ τουλάχιστον μια δήλωση της, είπα, της αρμόστριας και αν δεν μπορεί να παραστεί τις ε, χώρες που ασκεί την ε, Προεδρία και βεβαίως και στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Άρα λοιπόν θέλω να έχουμε όχι μόνο ε, δήλωση αλλά και συζήτηση και ψήφισμα για το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Σαλαφράνκα. Άρα αυτό ήταν η στήριξη της πρότασης αυτής. Είναι κάποιος κατά, όχι. Παρακαλώ λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν η δήλωση της Αντιπροέδρου και είπα της εκπροσώπου για την Λευκορωσία θα λάβει χώρα την Τετάρτη μετά τη συζήτηση για την Νιγηρία. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής προθεσμία. Απόψε 7 η ώρα για κοινά ψηφίσματα αύριο 7 η ώρα για τροπολογίες στα κοινά ψηφίσματα αύριο 8 η ώρα το βράδυ και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 15 Μαρτίου. Οπότε έχουμε κανονίσει την ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, κύριε Σπερώνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη διάσκεψη των Προέδρων είχα ζητήσει στην παρέμβαση της ε, Αντιπροέδρου, είπα της εκπροσώπου, ε, να γίνει αναφορά στην ε, ναυτική πειρατεία, κυρίως δε στους, ιδιαίτερη αναφορά στους Ιταλούς που κρατούνται ακόμα στην Ινδία. Δεν βλέπω όμως σε τέτοια αναφορά. Ελπίζω ότι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτό στη διάσκεψη των Προέδρων θα πραγματοποιηθεί. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνήσαμε να μην αλλάξουμε το τίτλο, να αναζητήσουμε από την κυρία Άστον να αναφερθεί στην μοίρα των δύο αυτών Ιταλών. Πράγματι έχουμε έρθει σε έπαφη μαζί της και έχει ενημερωθεί σχετικά. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίε και κύριοι, μου ζητήθηκε να κάνω μια δήλωση για το τσουνάμι και την καταστροφή στη Φουκουσίμα. και μετά τη δηλωσή μου θα ακολουθήσει συζήτηση με έναν γύρο από τον εκπρόσωπο της